Βεβαίως, εντάξει, αν θέλουμε και γραπτές απαντήσεις, ε, είναι δικαίωμά μα. Αλλά δεν είναι και πολύ ευγενικό την τελευταία μέρα, την τελευταία στιγμή, να τη πούμε ότι δεν σας δεχόμαστε. Εγώ προσωπικά έτσι το βλέπω, εντάξει. Ναι, η αρχική μου πρόταση ήταν να το αναφέρουμε απλά στην ε, συνάντηση, αλλά οι συντονιστές αποφάσισαν να έχουμε μια πιο έτσι στεναρή στάση και με ευρία πλειοψηφία. Αλλά μπορούμε, μπορούμε να αλλάξουμε, εσείς μπορείτε να αλλάξετε την ημερήσια διάταξη ως ε, σύνολο της Επιτροπής, έτσι. Πείτε το να ψηφίσουμε. Αν αποφασίσουμε όμως. Εντάξει, ωραία. Οπότε εγκρίθηκε η μερίσια διάταξη με αυτήν την τροποποίηση. Μετά. Τα πρακτικά έγκριση των πρακτικών της 6ης Νοεμβρίου και 20-21 Νοεμβρίου είναι στον φάκελό σας. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος συνεδρίασης εγκρίνονται. Επίσης υπάρχει η έκθεση της αποστολής μας στην Πολωνία 18 με 20 Σεπτεμβρίου. Μια άλλη ανακοίνωση αφορά τον κανονισμό για τα λοιπάσματα. Ένα πρώτος άτυπος τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί. Η ΙΜΚΟ είναι η αρμόδια επιτροπή, αλλά εμείς έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για τα θέματα των ρήπων. Οπότε έχουμε συμφωνήσει ότι η συγγήτρια της ΕΝΒΗ, η κυρία Γκαρδίνη, θα είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τους ρήπους. Έχουμε λοιπόν διερμηνία σε 21 γλώσσες, ε, ο φάκελος είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά και η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Κάτι το καινούριο έχουμε σήμερα. Η Γενική Διεύθυνση ITEC απέκτησε μια καινούρια κάμερα για ζωντανή μετάδοση βίντεο 360 μοιρών και θα την δοκιμάσουμε το απόγευμα στην ψηφοφορία. Μεταδίδονται συνήθως λοιπόν οι συνεδριάσεις μας, αλλά η κάμερα κοιτάει στον ομιλητή. Αυτή τη φορά θα έχουμε μετάδοση 360 μοιρών. Να το έχετε υπόψη. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με το πρώτο μας θέμα. Η Ευρωβινιέτα τέλη κυκλοφορίας ε, βαρέων οχημάτων για την χρήση υποδομών. Τον λόγο έχει λοιπόν ο εισηγητής, ο κύριος Ντάνς. Σας ευχαριστώ. Να σας ενημερώσω. Η Ευρωβινιέτα έχει κάπως λάθος όνομα γιατί περιέχει κάποιες προτάσεις για να φύγουμε ακριβώς από τις βινιέτες, τα αυτοκόλλητα των διοδίων. Τέλος πάντων έτσι λέγεται και έτσι θα την λέω και εγώ. Η οδηγία αυτή μας δίνει ένα νομικό πλαίσιο για την χρέωση τελών των φορτηγών για κάποιους δρόμους, ε, δηλαδή τα κύρια διευρωπαϊκά δίκτυα, δεν λέει πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν διόδια, αλλά αν γίνεται αυτό λέει το πώς θα πρέπει να γίνεται. Η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, και η αναθεώρηση της οδηγίας έχει στόχο να εφαρμοστεί καλύτερα η αρχή ο χρήστης και ο ρηπαίνων πληρώνει για να ισχύσει για όλα τα φορτηγά και σταδιακά και για τα γεωταχή και να αντικαταστήσει τις ε, βινιέτες με διόδια που θα αντικατοπτρίζουν την απόσταση. Να σας δώσω το πλαίσιο. Όταν μιλάμε για τα αέρια του θερμοκηπίου. Οι οδικές μεταφορές είναι υπεύθυνε για το 23% των εκπομπών και εξ αυτών το μεγαλύτερο κομμάτι βεβαίω προέρχεται από τα γεωταχή αλλά και τα φορτηγά αυξάνουν το μερίδιο τους. Το κόστος ε, αυτών των εκπομπών είναι ένα άλλο σημαντικό κόστος και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος ε, η ρήπανση αυτή είναι υπεύθυνη για πάνω από μισό εκατομμύριο θανάτους, ε, πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν μια αυξανόμενη ζήτηση για τις μεταφορές ε, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε και συμφόρηση στους δρόμους με ό,τι σημαίνει αυτό, καθυστερήσεις, σπατάλη καυσίμων και περαιτέρω εκπομπές. Όλα αυτά συμποσούνται σε 1 έως 2% του ΑΕΠ της Ένωσης. Σε γενικές γραμμές οι προτάσεις κομισιών είναι πολύ καλές, υποστηρίζω τις ε, προτάσεις τους και θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα χρέωσης ε, τελών για να μειωθούν οι εκπομπές και οι ρήποι. Αυτό γίνεται εφαρμόζοντας ε, καλύτερα την αρχή ο Ριπένων ε, πληρώνει και πρόθουμε έτσι και την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Η Κομισιόν ε, έχει προτείνει να επεκταθεί αυτό σε όλα τα βαρέα οχήματα και πουλμαν και λεωφορεία και τελικά και στα ελαφρά φορτίγα. Και το στηρίζω και το λέω γιατί και τα φορτηγάκια και τα πούλμαν και τα λεωφορεία παρά το ότι αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της ε, κυκλοφορίας και άρα της φθοράς ε, των υποδομών δεν πληρώνουν αναλογικά. Οπότε για να υπάρχει δικαιότερος ανταγωνισμός μεταξύ των μεταφορέων προτείνω να ισχύουν ε, αυτά και για τα μικρότερα φορτηγάκια, για την μεταφορά αγαθών που αυτή τη στιγμή έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ελαφρά φορτηγά οχήματα. Δηλαδή το όριο είναι οι 3,5 τόνοι. Τα μεγάλα φορτηγάκια χρησιμοποιούνται συχνά για την μεταφορά φορτίου ακριβώς για να παρακαμφθεί ο υφιστάμενος κανόνας και μάλλον θα συνεχιστεί αυτή η τάση. Όσον αφορά την χρέωση για τη χρήση των υποδομών, καλωσορίζω την πρόταση Κομισιόν για να καταργηθεί σταδιακά η βινιέτα γιατί δεν μας δείχνει ποια είναι η πραγματική χρήση του δρόμου. Κατ' ουσίαν δε η βινιέτα, η χρέωση κατά αποκοπή σε ενθαρρύνει να οδηγήσεις περισσότερο εφόσον είναι σταθερή η χρέωση. Έτσι, αν χρεώνουμε με βάση την απόσταση, θα έχουμε μια αναλογική χρέωση. Οπότε, για τα βαρέα οχήματα θα πρέπει να καταργηθεί μέχρι το 2022 και για τα ελαφρά οχήματα μέχρι το 2026. Ανέφερα μόνο το εξωτερικό κόστος, να αναφερθώ τώρα σε αυτό. Η πρόταση της Κομισιόν έχει στόχο να επεκτείνει την εξωτερική χρέωση η οποία αφορά την ρήπανση του αέρα και την ηχορύπανση και βεβαίως αυτό αφορά τα πιο επιβαρημένα τμήματα του οδικού δικτύου. Όμως το να το περιορίσουμε εκεί είναι και γραφειοκρατικό πρόβλημα. Εξάλλου η ρήπανση του αέρα μπορεί να ταξιδεύει εκατοντάδες χιλιόμετρα, οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια χρήση χρέωση των υποδομών για τα βαρέα και μη φορτηγά ε, από το 2021 και το 2026 αντιστοίχως. Τελικά θέλουμε να προωθήσουμε μια μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές και τα τέλη μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο για την υιοθέτηση αυτών των οχημάτων και για να επιταχύνουμε αυτήν την μετάβαση προτείνω να διατηρήσουμε την έκπτωση 75% για οχήματα μηδενικών εκπομπών που προτείνει η Κομισιόν. Προτείνω επίσης να διαγραφεί η εξαίρεση τεσσάρων ετών για τα πιο καινούργια οχήματα της πιο τελευταίας κλάσης Euro. Και έτσι νομίζω θα επιταχύνουμε την υιοθέτηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Τέλος, έχει σημασία ακριβώς να πηγαίνουν τα δύο αυτά στον συγκεκριμένο κλάδο για να το αποδεχτεί και η κοινωνία. Θα πρέπει δηλαδή έτσι να συντηρείται η σχετική υποδομή μειώνοντας και την ρήπανση και διευκολύνοντας την εισαγωγή οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Γιατί αν δεν βλέπει ο κόσμος που πάει τα λεφτά των δύο δύο, αν δεν υπάρχει σχέση με την συντήρηση των δρόμων, δύσκολα τα κράτη-μέλη θα τα δικαιολογήσουν. Αναμένω τη συνεργασία με τις άλλες ομάδες για να επιτύχουμε μια προοδευτική θέση που θα την αποστείλουμε στην Επιτροπή Μεταφορών. Καθώς είμαστε και εμείς συνδεδεμένη Επιτροπή για τα τέλη και την διακύμανσή τους σύμφωνα με τις εκπομπές και τους ρήπους. Σας ευχαριστώ. Στις 11 η ώρα θα έρθει εδώ ο κύριος Υπουργός, Υπουργός Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας. Οπότε προτείνω να έχουν περιορισμένο χρόνο οι ομιλητές. Λοιπόν, έχουμε τώρα τους κοιόδης. Ξεκινάω με τον κύριο Ζιπ. Ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό ας πούμε ο καθένας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι έχει προετοιμάσει μια πολύ ένα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο οδηγίας και πάει μάλιστα και προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως είπε και ο εισηγητής ο κύριος Ντάνς. Η ίσπραξη των ε, τελών των διοδίων ανά χιλιόμετρο αντί για τη βινιέτα που σχετίζεται με την διάρκεια χρήσης του α, οχήματος, ε, νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση. Σε ό,τι αφορά τώρα την, τον χρήστη των αυτοκινητοδρόμων, ίσως να είναι και πιο δίκαιο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, να είναι το σύστημα αυτό πιο δίκαιο. Παρ' όλα αυτά, το σύστημα της βινιέτας είναι αρκετά βολικό. Αγοράζει κανείς μια βινιέτα για κάποιο καιρό και το χρησιμοποιεί, τη χρησιμοποιεί όσες φορές θέλει μέσα σε αυτή την περίοδο για την οποία την αγόρασε. Βεβαίως πολλές φορές ακούμε ότι πρέπει κανείς να αγοράσει μια βινιέτα για, ένα, για ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη περίοδο ε, που ουσιαστικά ε, θα τη χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά ε, για να κάνει ένα μόνο ταξίδι. Και δεν αντικατοπτρίζει αυτό το χρόνο για τον οποίο έπρεπε να πληρώσουν την βινιέτα. Αυτό λοιπόν είναι αρκετά σημαντικό θέμα και σε ό,τι αφορά τις μεταφορές και σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Οι μεταφορές τους ή άλλως ε, συμβάλλουν σημαντικά στην ε, μόλυνση του αέρα. Και βεβαίως το θέμα των διοδίων είναι ένα θέμα πολιτικής. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη δεν ε, υποστηρίζαν ποτέ την επιβολή τέτοιων τελών και παρόλα αυτά τώρα σκέφτονται να επιβάλλουν τέτοιου είδους πληρωμές. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίσως ε, τους ε, αλλάξει άρδιν τα σχέδια. Οπότε καλό θα ήταν να το θυμόμαστε αυτό και να δούμε λίγο την κατάσταση ας πούμε στη Γερμανία. Νομίζω ότι ένα επίπεδο εναρμόνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλό θα ήταν. Το σύστημα αυτή τη στιγμή αλλάζει, τροποποιείται. Αυτό που πρέπει να ε, σκεφτούμε, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποιος θα είναι αυτός ο βαθμός εναρμόνισης. Εναρμονίζουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα τέλη. Ή εναρμονίζουμε και το πώς μπορούν να δαπανίσουν τα χρήματα που λέγουν τα κράτη-μέλη, εισπράττουν από αυτά τα διόδια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να πηγαίνουν σε σκοπούς σχετικούς με τις μεταφορές και βεβαίως να καλύπτουν και ε, περιβαλλοντικά κόστη. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούν κανέναν άλλον στόχο με αυτά τα χρήματα, τα κράτη-μέλη. Και επίσης θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς σχεδιάζει να περάσει από, την, από τις κατηγορίες ε, Euro στην προσέγγιση με τις ε, εκπομπέ άνθρακα. Και μάλιστα γιατί αυτές οι αλλαγές δεν έχουν μπει στο σχέδιο της οδηγίας. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που πρέπει να σας διακόψω. να ακούσουμε την κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη εγώ. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόταση. Ουσιαστικά, αν θεωρήσουμε ότι όντω υπάρχουν πολλέ εκπομπέ στου δρόμου και θέλουμε να τι αντιμετωπίσουμε, να τι διαχειριστούμε, θα πρέπει κανεί να πει να, ότι θα πρέπει να, καταγρα... να καταργηθούν τελείω τα τέλη αυτά και κάθε ένα να πληρώνει για την ε, ε μόλυνση που επιβάλλει χρησιμοποιώντα του δρόμου. Άρα ο, Ριπένον πληρώνει ε, σε πλήρη ε, ανάπτυξη. Επίσης, ε, πολλά καλά στοιχεία περιλαμβάνει η πρόταση. Ε, βεβαίως δεν μπορούμε να τα κάνουμε, να καταργήσουμε τα πάντα τώρα. Ε, το σύστημα θα ήταν να ε, δούμε κατά πόσο μπορούμε να απομακρυνθούμε σιγά σιγά έτσι ώστε να τα αφήσουμε να καταπέσουν τελικά τα παλιά συστήματα. Θα δούμε κατά πόσο η πρόταση αυτή είναι ρεαλιστική και κατά πόσο όντως μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα συνολικά το αν ε, μπορούμε να ζητήσουμε εξωτερικά κόστη και κάλυψη αυτών σωστό, το 75% για, τα, την έκπτωση να τη διατηρήσουμε επίσης σωστό. Ε, τώρα, αυτή την ε, πολιτική απελευθέρωση για τα, για τα τέλη για τις κατηγορίες Euro, ε, να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Είναι αρκετά φιλόδοξο ο στόχος και δεν ξέρω αν είναι ο σωστός τρόπος ωστόσο, αν θέλουμε δηλαδή να επιβραβεύσουμε κάποιον. Προφανώς κάθε, η, κάθε Υπουργός Οικονομίας χαίρεται όταν μπορεί να εισπράξει χρήματα. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν όντω ε, τα χρήματα αυτά που εισπράττονται χρησιμοποιούνται για θέματα μεταφορών και για θέματα επι, ε, ε, επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι προτάσεις της Κομισιόν πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και βεβαίως υποστηρίζω την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Ελπίζω ότι θα εκπνεύσει η οδηγία για την Ευρωβινιέτα και ελπίζω ότι όντως ο ε, Ριπένον θα ε, πληρώσει κάποια στιγμή. Βέβαια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή, αυτές τις αρνητικές πτυχές για το κλίμα και για το περιβάλλον, να τις αντιμετωπίσουμε μέσω των τελών χρήσης των φορτηγών για να κλείσουμε αυτά τα κενά που υπάρχουν. Η μελλοντική Ευρωβινιέτα και η σχετική ε, οδηγία θα πρέπει να επιφέρει ε, πρόοδο ό,τι αφορά την ε, αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Και βεβαίω θα πρέπει να επιφέρει και κάποια εναρμόνιση. Οι βλάβη στο περιβάλλον, οι κλιματικέ αλλαγέ θα πρέπει επίση να καλυφθούν ω θέματα μέσω τη οδηγία και οι ευαίσθητες γεωγραφικές περιοχές θα πρέπει να ε, τύχουν κάποιων ε, προτύπων προστασίας. Επίση, τα φορτικά κάτω των 12 ε, τόνων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δικέ μου θα έχουν στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκε εργασία και να αποφευχθεί το κοινωνικό dumping. Τα φορτικά σήμερα ταξιδεύουν από τι ανατολικές χώρες ε, και πραγματικά έχουν πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα από τους ε, οδηγούς ε, ιδιωτικών οχημάτων που είναι από τις δυτικές χώρες. Αυτά από μένα, Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ για τη δουλειά που έχεις κάνει. Νομίζω ότι έκανε ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή. Ε, νομίζω ότι περίπου 60% της ε, μόλυνσης προκύπτει από τα επιβατικά οχήματα. Και βεβαίως θα πρέπει και τα υπόλοιπα είδη οχημάτων να ε, εντάσσονται σε αυτή την πρόταση. Βεβαίως πρέπει να δούμε την ε, χρέωση ανά απόσταση, ανά χιλιόμετρο και να ε, δώσουμε κίνητρα για να είναι πιο αποτελεσματικά και πιο καθαρά τα ταξίδια μας με τα οχήματα. Ε, η, επίσης η ανάγκη για μηδενικές εκπομπές επίσης είναι άμεση και αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για την μόλυνση του περιβάλλοντος. Και επίσης θα πρέπει να δούμε και, άλλους, και άλλες επιμολυντικές ουσίες οι οποίε έχουν μεγάλο αντίκτυπο και στην υγεία και αυτό το εργαλείο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το μέσο των μεταφορών θα πρέπει να αρχίσει να πληρώνει το μερίδιο που το αναλογεί. Το ελάχιστο εξωτερικό κόστος βεβαίω θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλο το δίκτυο, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ τρόπων μεταφορών. Και για να το ε, επιτείνουμε αυτό, το 100% των ε, ε, των αυτοκινητοδρόμων καλύπτεται από, διό, από διόδια. Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισοτιμία όπλων για όλους τους εμπλεκόμενους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον ΣΕΜΠ, για την πρόταση που υπέβαλε για να υποβάλει αυτή τη νέα πρόταση της Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι πεπισμένος ότι η πρόταση αυτή της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, ε, τονίζει την απαράβατη αρχή ο πληρώνει». κληρώνει. Ως προς άλλους τομείς ε, είμαι υπέρ των βασικών τελών της Επιτροπής και της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής αυτής της οδηγίας για να μην περιλαμβάνει μόνο τα βαρέα αλλά και τα ελαφρά οχήματα με βάση τη διάρκεια δικαιωμάτων και χρήσης. Αλλά ε, θα πρέπει αντίθετα να περάσουμε στην αρχή της χρήσης, της χρονοχρήσης. Γι' αυτό αυτή η γνωμοδότηση νομοθετικού περιεχομένου θα πρέπει να έχει ένα ρεαλιστικό πλαίσιο καθώς και φιλόδοξο με τον ορίζοντα του 2020, δηλαδή την ε, ανάληψη του κόστους λαμβάνοντας υπόψη την ε, ρήπανση και ιδιαίτερα την ηχορύπανση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εσωτερήκευση του κόστους έτσι ώστε στη συνέχεια να επενδυθούν αυτά τα τέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική κάλυψη των ε, εξόδων και τα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για επενδύσεις, έτσι ε, ώστε να ξεπεράσουμε το μοντέλο που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα. Η κυρία Μελέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αυτό το θέμα θέτει ορισμένα ζητήματα για μας. Για τον τρόπο δηλαδή τελών των ε, εθνικών οχημάτων και εκείνων που προέρχονται από το εξωτερικό είναι γεγονός ότι μία χώρα διέλευσης όπως η Γαλλία θα πρέπει να καλύψει τη ρήπανση καθώς ε, και τη συντήρηση των ε, οδικών δικτύων για τα εθνικά και μη οχήματα. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί Για πρώτη φορά μιλάμε για μια ευρωπαϊκή επιβολή τελών και θα ε, επαγρυπνούμε ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Η έκθεση πάει στη σωστή κατεύθυνση. Δύο-τρία πράγματα θέλω να πω απλώ. Ιδιαίτερο σωστό είναι να, τα μικρά οχήματα να τα συμπεριλάβουμε στο όλο σύστημα αυτό των διοδίων. Όλο και περισσότερα οχήματα βρίσκονται στους αυτοκινητοδρόμους αυτό δεν είναι όμως θέμα διοδίων. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα της ξεκούρασης και των ε, ε, διαστημάτων οδήγησης. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχουν ανεξάρτητα διόδια, διόδια να δώσουμε και μια μετάβαση μέχρι το 2025 για τα φορτηγά. Βεβαίως κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να συμπεριλάβει νέες βινιέτες μέχρι τότε στο σύστημα. Δεν θέλουμε να επιδεινώσουμε ακόμη περισσότερο την τρέχουσα κατάσταση. Τώρα, για, τον, για τη στοχοθέτηση, νομίζω ότι είναι σωστή μεν, αλλά θα πρέπει να τη δομήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε ο, ο πληθυσμός που ζει κοντά στις, ε, στους αυτοκινητοδρόμους να, βελτιώσει, να βελτιώσει τους, ε, την ποιότητα ζωής του. Να μην ξεχνάμε ότι πολλοί αυτοκινητόδρομοι αντιμετωπίζουν πολλά ε, προβλήματα και ταυτόχρονα είναι και πολύ σημαντικές ε, πηγές εσόδων. Οι υποδομές σίγουρα μπορούν να βελτιωθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν και οι συνθήκες ζωής των πολιτών που ζουν κοντά σε τέτοιους δρόμους. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. thank you. Um, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Η Επιτροπή καλωσορίζει τις προτινόμενες τροπολογίες και γνωρίζουμε ότι η έκθεση συμβαδίζει με την έκθεση της κυρίας Ρεβονταλόν στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα λάβουμε υπόψη τα μέτρα που προτείνονται και σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, η αντικατάσταση των ε, αξιών αναφοράς με, ελάχιστες, ε, με ελάχιστα όρια. Επίσης, θα προωθήσουμε τις, ε, τις προθεσμίες σε σχέση με την απαλυφή αυτών των όριων σταδιακά προτείνουμε, δεχόμαστε μάλλον και τις προτινόμενες αλλαγές για τα οχήματα που εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή ένα 75% θα μπορούσε να ισχύσει ήδη από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό το 75% όσο αφορά το earmarking. Ξέρετε ότι η Επιτροπή είχε υποστηρίξει την χρήση των διαδίων για τις νέες επενδύσεις στον τομέα μεταφορών, έτσι ώστε να γίνει πιο βιώσιμος ο τομέας μεταφορών. Γι' αυτό δεχόμαστε και τα, το επιπρόσθετο σημείο στο άρθρο 9 της οδηγίας για να δώσουμε κίνητρα για την χρήση αυτών των εσόδων για καθαρές μεταφορές. Ε, και θα ήθελα να προσέξετε και το εξής. Ορισμένα άλλα στοιχεία που υπάρχουν στην οδηγία που ενέχονται σε αυτό το άρθρο αφορούν την ασφάλεια των οδικών μεταφορών και την στάθμευση. Αυτά έχουν μεταφερθεί αλλού και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη εκ νέου. Όσον αφορά την ε, διακύμανση τελών σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίων του άνθρακα, δεν έχουν οριστεί οι προδιαγραφές επακριβώς στην οδηγία, γιατί τα αναγκαία στοιχεία εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για βαρέα οχήματα δεν είναι διαθέσιμα ακόμα. Τα ετοιμάζουμε και τα υπολογίζουμε. Έχουμε δώσει τελική μορφή στη μεθοδολογία μας και τη στιγμή που υπάρχουν επιστοποιημένα στοιχεία για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα τότε θα μπορούσαμε να προβάλλουμε ένα πρότυπο διαφοροποίησης ανακλάση οχημάτων και σύμφωνα με τις εκπομπές. Θα το δούμε λοιπόν σε μια κατεξιοδότηση πράξη και βεβαίως υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα. Κατά πόσο δηλαδή το Κοινοβούλιο θα ήθελε και τα κράτη-μέλη θα ήθελαν να δεχτούν τις κατηξουσιοδότηση πράξεις. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε διαφοροποιημένα τέλη ανάλογα με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα βραχυπρόθεσμα παρά να περιμένουμε για την πλήρη αλλαγή της οδηγίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντάνς να απαντήσει εντάχει. Ναι, θα είμαι σύντομος. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας και την Κομισιόν. Συμφωνούμε όλοι νομίζω στις γενικές αρχές. Ε, εντάξει, υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των ομάδων, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τίποτα το οποίο δεν ε, λύνεται. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη στήριξης ε, των αρχών της πρότασης αυτής αλλά και μια αναθεώρηση του συστήματος δύο-διών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες που θα εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, ακόμα και αν φύγουν. Ονόματα δεν λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνω στην ώρα λοιπόν. Προθεσμή για απολογίες 1 Φεβρουαρίου. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή 26-27 Μαρτίου. Και Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Νομοντήμο, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ιδάτων της Βουλγαρίας. Κάποιος πρέπει όμως να φέρει τον κύριο Υπουργό. Uh, Καλημέρα, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Καλώς ορίζω τον κύριο Δήμοφ, Υπουργό Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας. Συγχαίρω και την Βουλγαρία για την πρώτη της Προεδρία και σας εύχομαι καλή επιτυχία τους επόμενους έξι μήνες ως συνήθως. Λοιπόν, στην αρχή της Προεδρίας ε, έρχεται ο Υπουργός, παρουσιάζει τις προτεραιότητες ε, στο θέματα περιβάλλοντος, ε, κλίματος και θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων βεβαίως με τα μέλη της Επιτροπής μας. Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι ο Υπουργός θα καλύψει τα ζητήματα ασφάλειας τροφίμων που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Αναμένουμε λοιπόν την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω την μητρική μου. Αλλά Αν δεν αρκεί η μία μισή ώρα μπορούμε να συνεχίσουμε μετά με ερωτήσεις. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσω βουλγαρικά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα να αναφέρω το πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας με τα μέλη της Επιτροπής για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας ε, στο περιβάλλον. Ως ε, ένα από τα παλαιότερα κράτη της Ευρώπης, ε, βεβαίως η Βουλγαρία συνεισφέρει στην πολιτισμική ταυτότητα της Ευρώπης λόγω της της ιστορίας της και των επιδευμάτων της ε, στην, ε, στις τέχνες και βεβαίως δώσαμε στην Ευρώπη ένα από τα τρία αλφαβητά της, ε, το κυριλικό. Η Βουλγαρία έχει υποστεί πολλές εισβολές επί αιών, με πολλές θυσίε και εξακολουθούμε να είμαστε ο φύλακας της νοτιοανατολικής πύλης της Ευρώπης και σήμερα. Και ως φύλακας θα έλεγα ο ρόλος μας αυτός εκτείνεται και στο θέμα του φυσικού περιβάλλοντος. Έχουμε πολύ μεγάλη βιοπικιλότητα στην Βουλγαρία και σε σχέση με αυτό ε, εξετάζουμε βεβαίως και την οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο του ε, πώς θα επιτύχουμε μία ισορροπία με το περιβάλλον και ακριβώς ε, προς αυτή την κατεύθυνση τα έργα του Προεδρία ως Προεδρία του Συμβουλίου. Έχει μεγάλη σημασία για εμάς ε, να ξεκινήσουμε έναν αποτελεσματικό και ανοιχτό διάλογο με το Κοινοβούλιο που είναι συνομοθέτης ε, και θεωρώ ότι όλα αυτά είναι σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποδεχόμαστε βεβαίω την πρόκληση αυτή της πρώτης βουλγαρικής προεδρίας και θα ήθελα εδώ πέρα να επιβεβαιώσω την ε, σταθερή μας τοποθέτηση υπέρ ενός διαλόγου για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και τις βασικές ε, ευρωπαϊκές αξίες. Η Ευρώπη και οι πολίτες της χρειάζονται περισσότερη ασφάλεια, σταθερότητα και αλληλεγγύη. Η ασφάλεια σημαίνει εδώ πέρα να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη υγεία και την υγεία του πλανήτη, σταθερότητα, δηλαδή να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας και βεβαίως εστιάζοντας προς τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Αλληλεγγύη, βασιζόμενη στην συνοχή και την σύγκληση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις ε, κοινωνικο-οικονομικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Εξετάζουμε λοιπόν ε, τα αποτελέσματα της ε, κυκλικής οικονομίας και θα εργαστούμε για να δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και ένα φιλικό περιβάλλον για καινοτόμες λύσεις. Η βασική μας προτεραιότητα είναι η κυκλική οικονομία και η οικοκαινοτομία καλωσορίζουμε το μίνι πακέτο που ενέκρινε η Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά την κυκλική οικονομία. Σκοπεύουμε να δώσουμε προτεραιότητα στην στρατηγική για τα πλαστικά και θα οργανώσουμε μια υπουργική διάσκεψη τον Μάρτιο. Θα εστιάσουμε την συζήτηση στο πώς θα αυξηθεί η ανακύκλωση και θα μειωθεί η απανθράκωση και οι χωματερέ. Επίσης, σκοπεύουμε να ευθύσουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Ιούνιο. Τα συμπεράσματα αυτά θα αποτελέσουν κατευθυντήριε γραμμέ για την Κομισιόν για τα επόμενα βήματα και μέτρα της στρατηγική που θα πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα και κατά προτεραιότητα. Και εδώ θα ήθελα να πω πως η συζήτηση θα περιλαμβάνει και ανακοίνωση για το πώς ακριβώς ε, θα συνδυάζονται τα νομοθετήματα περί χημικών και αποβλήτων. Βεβαίω έχουμε και το θέμα της ποιότητας του αέρα που είναι ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα και έχουμε έτσι τα θέματα ακριβώς της μείωσης ε, του αντικτύπου των ρήπων. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζουν μόνο τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη 16 κρατημέλη σύμφωνα με αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Γι' αυτό θα εστιάσουμε τις ε, προσπάθειές μας ε, για να χρησιμοποιήσουμε διαφορούς μηχανισμούς ε, και καινοτόμες λύσεις για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα και να γίνουν πιο δημοφιλείς αυτοί οι μηχανισμοί για να προστατεύσουμε την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και το περιβάλλον. Αυτό θα είναι και το βασικό θέμα της διάσκεψης για την οικοκαινοτομία που οργανώνουμε στις 5 και 6 Φεβρουαρίου μαζί με την Κομισιόν στη Σόφια. Η ποιότητα του αέρα επίσης θα συζητηθεί ως θέμα στο άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος ε, τον Απρίλιο. Και δράτω με τις ευκαιρίες κυρία Πρόεδρε να σας προσκαλέσω και στις δύο αυτές εκδηλώσεις. Προτεραιότητά μας επίσης είναι το θέμα της καλύτερης νομοθεσίας με στόχο την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής ε, νομοθεσίας. Είναι κοινή μας ευθύνη αυτό, καθώς ε, η τρέχουσα, η φυστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, περιέχει κάποια αντιφατικά στοιχεία χωρίς σειρά προτεραιότητας και έτσι υπάρχει, δεν υπάρχει η απαραίτητη νομική προβλεψιμότητα. Και βεβαίως υπάρχει αφενός η περιβαλλοντική νομοθεσία και η νομοθεσία γεωργίας, ενέργειας και κλίματος από την άλλη. Και πρέπει ακριβώς να ξεπεράσουμε αυτές τις αντιφάσεις για να αγγιθούμε την καλύτερη εφαρμογή και να επιτύχουμε ε, τους στόχους μας. Οπότε, πέρα από το άτυπο συμβούλιο του Απριλίου, θα δούμε το ζήτημα στο πλαίσιο του πρασινίσματος στην ε, υπουργική διάσκεψη του Μαρτίου. Και τέλος για να μην υπάρχουν παρερμηνίες θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχει πολιτική συνένεση στην Ευρώπη για τα ζητήματα πολιτικής αλλαγής και τα σχετικά μέτρα. Και η Βουλγαρία είναι το τμήμα αυτής της ε, συνένεσης. βεβαίως ε, προετοιμαζόμαστε και για την 24η ε, διάσκεψη των μερών για την κλιματική αλλαγή, για την επικαιροποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων. Θα δούμε έτσι τα ζητήματα προσαρμογής ε, στην κλιματική αλλαγή όσον αφορά το τι μπορεί να γίνει στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της Ένωσης. Το άλλο νομικό πλαίσιο που αφορά τις μεταφορές χωρίς εκπομπές είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Θα κοιτάξουμε τις σχετικές διαπραγματεύσεις για την πρόταση για τα νέα βαρέα οχήματα, την παρακολούθηση και τις αναφορές. Έχουμε ξεκινήσει εντατικές συζητήσεις ε, επί της σχετικής πρότασης ε, για τις προδιαγραφές εκπομπών για νέα οχήματα, αυτοκίνητα και φορτηγά είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, τους πολίτες και την αυτοκινητοβιομηχανία. Θα οργανώσουμε μία συζήτηση σε επίπεδο υπουργών τον Ιούνια για το θέμα αυτό. Συνοψίζοντας, η Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δει κάποιες προκλήσεις που δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε και να φανταστούμε εύκολα. Κρίσεις που είχαμε ξεχάσει σε καιρούς ε, εφημερίας. Θεωρώ ότι οι προκλήσεις μας ενώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και η κρίση μας διδάξει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσουμε στην κρίση αυτή με περισσότερη Ευρώπη, γιατί το μέλλον ανήκει σε μια Ευρώπη ενότητας, ευημερίας και αλληλεγγύης. Η ισχύ είναι τη λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να ακούσουμε τους συντονιστές πρώτα των πολιτικών ομάδων για να θέσουν τα ερωτήματά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Λαβία πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, για την παρουσία σας σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και για τα θέματα τα οποία ορίσατε ως προτεραιότητα της Βουλγαρικής Προεδρίας. Έχει μεγάλη σημασία ε, η συνεργασία μεταξύ των δύο συνομοθετών του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας ορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματός μας. Μιλήσατε για την σημασία ορισμένων νομοθετικών πακέτων που το Συμβούλιο θα εφαρμόσει μέσα στα πλαίσια της εξάμηνης Προεδρίας, ξεκινώντας από την ε, κυκλική οικονομία, ανακύκλωση και ούτω καθεξής. Βεβαίως ε, συμμεριζόμαστε αυτούς τους στόχους όπως ορίστηκαν από την προηγούμενη Προεδρία για να περάσουμε στην εφαρμογή και να θέσουμε σε εφαρμογή και αυτό το νομοθετικό πλαίσιο με την λήξη της Προεδρίας τον Ιούλιο ως προς την προστασία των πολιτών, το περιβάλλον, το πρασίνισμα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Είναι θέματα που απασχολούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος, ιδιαίτερα ως προς την ΚΑΠ, που οδηγείται σε μια επανεθνικοποίηση και μία ε, αντιμετώπιση, επιμέρους αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Σε σχέση με την επόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό, είχε προβλεφθεί ότι το 2015 η Επιτροπή θα είχε επανεξετάσει το παράρτημα 1 σε σχέση με την ποιότητα των ε, υδάτων, αλλά δεν επικαιροποιήθηκε αυτό το παράρτημα. Εκεί γίνεται μνήα για το πόσιμο νερό και τη σύσταση του νερού και από όσο γνωρίζουμε ίσως υπάρξουν διακρίσεις αυτής της πολύτιμης πηγής και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζουν ένα όριο 2,4 ε, χιλιόγραμμα, ενώ εμείς μιλάμε για περιεκτικότητα ενός χιλιογράμμου. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε το παράρτημα της οδηγίας για να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή, διότι το, το νερό είναι μια πολύτιμη πηγή και θα ήθελα τη δική σας γνώμη επί του θέματος. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Καταρχήν να σας συγχαρώ για το εξάμεινό σας και γιατί είναι το πρώτο εξάμεινο υπό Βουλγαρική Προεδρία. Έχετε πολύ σημαντικά νομοθετικά ζητήματα. Σας περιμένει πολύ μεγάλη εργασία σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στα οχήματα, αλλά αυτό αφορά και τα βαρέα και ελαφρά οχήματα. Πρόκειται για σημαντικούς στόχους για να φτάσουμε στα ε, αποτελέσματα και συμπεράσματα της Συμφωνίας των Παρισίων και για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Επίσης μιλήσατε για την ε, κυκλική οικονομία και την ε, χρήση των πλαστικών. Ως προς την κυκλική οικονομία, μιλήσατε για μία πρώτη σας προτεραιότητα. Εγώ ήμουν η συγγήτρια επί του θέματος και φτάσαμε σε μια προσωρινή συμφωνία τον προηγούμενο μήνα μετά από μια δυσχερή διαπραγμάτευση. Δυστυχώς έχει ε, σταματήσει αυτό το θέμα στη γραμματεία του Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να το προωθήσετε έτσι ώστε να, ώστε να τηρηθεί αυτό το πλαίσιο και να τηρήσουμε και τις ε, προδιαγραφές ως προς την ανακύκλωση και τα απόβλητα. Μιλήσατε και για την ανάπτυξη της ε, καινοτομίας και θα πρέπει να μιλήσουμε για οικοκαινοτομία για ολόκληρο τον κύκλο ζωής και για να θέσουμε σε εφαρμογή τη νέα οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν την πρόταση για την κυκλική οικονομία. Αλλά αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα της ανάπτυξης και να φτάσουμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη πριν από τους άλλους για ανταγωνιστικούς λόγους, δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για το περιβάλλον και το είπατε εσείς, θα πρέπει να προωθήσουμε μια οικονομία που να προστατεύει το περιβάλλον. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα φτάσετε σε ένα κοινό έγγραφο με το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας γιατί μιλάμε όχι μόνο για περιβάλλον αλλά και βιώσιμη οικονομία. Σας υπενθυμίζω ότι έχετε δύο λεπτά ο καθένας. Η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την, τον Υπουργό και θα ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα που δεν βρίσκεται στη νομοθετική ατζέντα, αλλά που είναι ύψη της ε, σημασίας. Πιστεύω ότι αυτό που μετρά για το κοινό μας είναι η ποιότητα του αέρα είδα τις εκθέσεις των περιφαλλοντικών οργανώσεων για τη Βουλγαρία και είδαμε πώς έχει η κατάσταση και για τη Βουλγαρία. Θα ήθελα να αναλυφθεί δράση χωρίς να περιμένουμε νομοθέτηση, δηλαδή κάποια δήλωση προθέσεων από τα κράτη-μέλη ότι είναι δια τεθειμένα να αναλάβουν μέτρα για την ποιότητα του αέρα. Και με τα νέα της Επιτροπής βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν μακρύ κατάλογο παραβιάσεων από τα κράτη-μέλη. Φτάσαμε σε ένα κρίσιμο σημείο και δεν ξέρω κατά πόσο η δική σας Προεδρία θα μπορούσε να αναλάβει δράση. Με βάση την εθνική σας εμπειρία, τι θεωρείτε ότι μπορείτε να προωθήσετε. Ε, ο κύριος Κερμπράντη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Υπουργό Ντίμοφ που είναι εδώ μαζί μας. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Μιλήσατε για συνένεση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη Βουλγαρική Προεδρία για τις κλιματικές αλλαγές, αλλά φαίνεται να βάζετε ορισμένα ερωτηματικά κατά πόσο δηλαδή το είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα και αυτό αφορά και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Επειδή θα είσαστε επικεφαλής πολλών συνεδριάσεων για τις κλιματικές αλλαγές, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η προσωπική σας θέση επί του θέματος. Ως προς την ποιότητα του αέρα, χαίρομαι γιατί είναι μια άμεση προτεραιότητά σας, αλλά είσαστε μαζί με την Πολωνία και αμφισβητείτε μία νομοθεσία που έχει ήδη εγκριθεί για τα νέα όρια καύσης, ε, τα νέα όρια για τα μεγάλα εργοστάσια ή μονάδες καύσης. Μπορείτε να μας πείτε ποια θα είναι η προτεραιότητά σας τη στιγμή που έχετε καταγγείλει νομικά αυτές τις νέες ε, προδιαγραφές. Επίσης, ως προς την βιοπικιλότητα, για το 2020 βλέπω ότι ε, δεν υπάρχει τίποτα που να εντάσσεται στο πρόγραμμά σας. Αν θέλουμε όμως να βρεθούμε πιο κοντά στους στόχους βιοπικιλότητας για το 2020, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση Γι' αυτό δεν ξέρω κατά πόσο η Βουλγαρική Προεδρία προτίθεται να κάνει κάτι στον τομέα της βιοποικιλότητας για να σώσει την φύση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω ότι η κυκλική οικονομία και η νομοθεσία για τα απόβλητα είναι πολύ σημαντικά θέματα Παρ' όλα αυτά έχουμε άλλο ένα πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε την, στην προηγούμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο για το κλίμα και περιλαμβάνει τρία έγγραφα, ΛΟΛΟΣΙΕΦ, διακυβέρνηση και βιοκαύσιμα. Και επίσης ε, ενεργειακή επάρκεια αυτά δεν τα αναφέρατε, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε σκοπό να προωθήσετε και τα θέματα αυτά, είτε μέσω άμεσης εφαρμογής των εκθέσεων και των ε, νομοθετικών πράξεων, είτε με τη μορφή τριμερών διαλόγων. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εσάς τους τριμερείς διαλόγους. Και επίσης, ε, κάτι για τα βιοκαύσιμα. Ποια είναι η άποψή σας για το phase-out της πρώτης γενιάς βιοκαυσίμων εντός μιας πολύ σύντομης προθεσμίας και, τα βιοκαύσιμα, και την κατάργηση των βιοκαυσίμων από φινικέλαιο που θέλουμε να αντικατασταθούν από το 2020 και μετά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μελάν. Α, δεν είναι εδώ. Άρα κλείνουμε τον πρώτο γύρο ερωτημάτων προς τον Υπουργό και θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικά τα ερωτήματα που μου θέσατε. και βεβαίως θα μπορέσω να σας δώσω αρκετές προφορίες. Ε, μου είπατε ότι στην ε, πρώτη μου παρέμβαση έπρεπε να είμαι αρκετά σύντομος και γι' αυτό δεν μπορούσα να σας αναφέρω τα πάντα. Έτσι, μερικώς απαντώ σε ένα σχετικό ερώτημα. Να αρχίσω από την αρχή λοιπόν. Ε, κύριε Λαβία, Βεβαίω ότι σχετίζεται με την υγεία των πολιτών, με τη δημοσία υγεία μας απασχολεί. Τόνισα την ατμοσφαιρική ρήπανση, την ποιότητα του αέρα, αλλά δεν ε, σημαίνει αυτό ότι δεν είναι σημαντικό το περιβάλλον, η γενικότερη ρήπανση και άλλα τέτοια θέματα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι στην ε, Βουλγαρία έχουμε ε, από τα πιο υψηλής ποιότητας πόσιμα νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν θέλω να πάρω τώρα την, ε, το ρόλο του εθνικού εκπροσώπου. Τα αποτελέσματα της οδηγίας για το πόσιμο νερό δείχνουν ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι ένα από τα σημεία κλειδιά για την επίτευξη μιας υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, μέσω αυτής της αναθεώρησης, ε, καταγράφηκαν και κάποιοι ε, προβληματικοί τομεί, οι οποίοι χρειάζονται βελτίωση. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την παροχή πληροφοριών στους πολίτες για τα πρότυπα εξασφάλιση ποιότητας. Οπότε περιμένουμε την σχετική πρόταση της ε, Κομισιόν για να αναθεωρήσουμε την οδηγία έτσι ώστε να καλύψουμε και αυτά τα εκρεμή θέματα. Σίγουρα θα έχουμε μια οδηγία η οποία θα εξασφαλίζει ένα ισότιμο επίπεδο προστασίας ε, από την ε, μόλυνση των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φυσικά καταλαβαίνουμε τη σημασία, αλλά βεβαίω για να μπορέσουμε να δράσουμε περιμένουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Μποναφέ, θέσατε διάφορα σημαντικά ερωτήματα για την κυκλική οικονομία, για την οικοκαινοτομία και την ανάπτυξη. Να ξεκινήσουμε την κυκλική οικονομία. το περιβάλλον είναι πραγματικά το καταλληλότερο παράδειγμα κυκλική οικονομίας. Πρέπει από το περιβάλλον να μάθουμε πώς να δημιουργήσουμε μια κυκλική οικονομία. Η οικοκοινοτομία φυσικά είναι σημαντική για το τρίο των προεδριών, γιατί πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κρίσεις. Και νομίζω ότι η δυνατότητα να εφευρίσκουμε μας βοήθησε να αναπτυχθούμε. Και νομίζω ότι ε, αυτή τη φλόγα της ε, ευρωπαϊκής διάνοιας θα πρέπει να την καλλιεργήσουμε περαιτέρω. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή που κατά πάσα πιθανότητα θα κρατήσει και πέραν της δικής μας Προεδρίας, αλλά σίγουρα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση και κατά τη διάρκεια των επόμενων Προεδριών. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εντό έξι μηνών ή ενό χρόνου ακόμα να λύσουμε το θέμα αυτό. Είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να προωθήσουμε, να διευκολύνουμε. Τώρα το πακέτο για τα απόβλητα. Η Ιστονία και η Ιστονική Προεδρία πραγματικά έκανε πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τα απόβλητα. Οπότε τον Φεβρουάριο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε στην Κορεπέρ το πακέτο αυτό, έτσι ώστε να πάρει το δρόμο του. Επίσης, α, ακούστηκαν κάποια σχόλια για την ποιότητα του αέρα. πρέπει να ληφθούν μέτρα, βεβαίως. Ισχύει αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω μιας νομοθετικής πράξης, είτε και όχι. Υπάρχει ένας ε, χάρτης που έρχεται από την ε, EEA, που δείχνει τις ψηλότερες ε, θερμοκρασίες Αυτό δεν το έχουμε προχωρήσει ακόμη, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προωθήσουμε κυρίως την, ε, την ε, ε, πρωτοβουλία αυτή για τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία είναι στην Ευρώπη αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε και οι πολίτες τους να θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι όντως το σπίτι τους. Όταν λοιπόν μιλούμε για συγκεκριμένα μέτρα, θα ήθελα να συμπεριληφθούν σε αυτά και τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχω καλέσει τους Υπουργούς ε, ε, Περιβάλλοντος των Δυτικών Βαλκανίων να ε, παραστούν στην Σύνοδο στη Σόφια στις 5 και 6 Φεβρουαρίου, όπου θα συζητήσουμε τα θέματα οικοκαινοτομίας και της ποιότητας του αέρα. Οπότε η, μέσω της οικοκαινοτομίας θέλουμε να προωθήσουμε και την βελτίωση της ποιότητας του αέρα και ελπίζουμε ότι θα συμπεριλάβουμε στο διάλογο αυτό και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων γιατί ξέρετε ότι ο αέρας δεν έχει σύνορα και είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλους τους Ευρωπαίους. Ο κύριος Γερμπράντι έθεσε διάφορα ζητήματα. Όπως είπα στην αρχή, μπορώ να θέσω διάφορα ερωτήματα που απευθύνονται σε μένα προσωπικά, αλλά εγώ είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της Βουλγαρικής Προεδρίας, εκπρόσωπος του ε, Συμβουλίου αυτή τη στιγμή. Οπότε η προσωπική συζήτηση που θέλετε να κάνουμε μπορεί να γίνει εκτός αυτής της αίθουσα και ευχαρίστω να την κάνουμε. Στην ε, παρέμβαση μου είπα ότι υπάρχει η πολιτική ε, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαίως η επιστήμη πάντα ψάχνει. Γι' αυτό δίνει πάντα περαιτέρω επιχειρήματα για να καταλήξουν οι πολιτικοί σε μια συμφωνία. Και μετά αυτή η συμφωνία να μεταφραστεί σε μέτρα, σε πράξεις. Και γι' αυτό το ανέφερα στην αρχική μου παρέμβαση. Επίσης, Είπατε ότι η ε, Βουλγαρία μαζί με την Πολωνία αντιτίθεται σε μία ε, δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η ποιότητα του αέρα είναι πρωτοβουλία, πρωτο, Βουλεία της ε, Βουλγαρίας και άλλων 16 χωρών. Αυτό δεν αντιτίθεται στο γεγονός ότι όντως είμαστε αντίθετοι με μία πράξη σε σχέση με, τον, με τη νομική διαδικασία και το πώς υιοθετήθηκε η νομοθεσία. Φυσικά θα πρέπει να παρακολουθείτε. Χρειαζόμαστε και κάποιες δυνατότητες να παρεμβαίνουμε. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθηθεί η δράση αυτή. Αν τώρα το δικαστήριο μας δώσει δίκιο, εντάξει. Αν δεν μας δώσει δίκιο, πάλι εντάξει. Το κράτος δικαίου όμως είναι μία από τις βασικές αξίες και θεωρούμε ότι έχουμε δικαίωμα να είμαστε αντίθετοι με μία νομοθετική πράξη και γι' αυτό από κοινού υποβάλλουμε το έτοιμο αυτό με την Πολωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα την προστασία της φύσης. Εμείς ε, είμαστε μία από τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό περιοχών Natura 2000. Πάνω από 35% της ε, επικράτειας χώρας μας καλύπτεται και Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να υπάρξει και σεβασμό στο περιβάλλον, στην διατήρηση τη βιοπικιλότητα. Είναι σημαντικό αυτό φυσικά και για την οικονομία. Να προστατεύσουμε το περιβάλλον Επίση είναι σημαντικό ώστε να μπορούν να ζουν σε σωστέ συνθήκε. Οι πολίτε δεν μπορεί να προωθήσει κανεί είτε τη μία πλευρά είτε την άλλη. Μόνο μέσω ε, ισότιμης όλων αυτών των πτυχών θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι πολίτε να απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα ζωή. Για τα θέματα της ενέργειας, νομίζω ότι προσπάθησα και στην αρχή να τα θίξω και βεβαίως έχουμε και τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση. και την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Βουλγαρική Προεδρία βεβαίως θα, θα συνεχίσει τη δουλειά πάνω στο πακέτο για την καθαρή ενέργεια βασιζόμενοι στα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της Εστονικής Προεδρίας. Η Βουλγαρική Προεδρία επίσης περιμένει να ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι για τον ε, κανονισμό για τη διακυβέρνηση και επίσης το σχέδιο οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περιμένουμε ε, εντατικές ε, και καρποφόρες συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι όλοι θα είμαστε και διαφανείς και αποτελεσματικοί. Και εδώ θέλω να υπογραμμίσω κάτι. Όλοι σας αντι εκπροσωπείτε τα, τα, διάφορα συμφέροντα των πολιτών σας, των εκλογικών σας περιφερειών, οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των συμφερόντων. Και εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ 28 κρατημέλη, οπότε πρέπει να φροντίσω και τα δικά του συμφέροντα. Η κοινή δουλειά λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι ιδιαίτερο σημαντική για να μπορέσουμε να εξεύρουμε αυτή την ισορροπία, ισορροπία δηλαδή με τα κρατημέλη και από την άλλη ισορροπία των ε, ψηφοφόρων σας. Οπότε η δική μας η πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή για να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Παρακαλώ να μην μακρηγορείτε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μία από τις προτεραιότητες σας είναι τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως είπατε, και η ένταξή τους. Υπάρχει ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, ε, ιδιαίτερο, που μπορεί να είναι και αρμοδιότητός σας. Πριν από ένα μήνα, και όχι για πρώτη φορά, είχαμε τεράστια οικολογική καταστροφή στην θάλασσα προερχόμενοι από τους ε, γείτονές μας. Ε, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η πόλη μου, το Ντουμπρόβνικ, απειλείται από την οικολογική αυτή, οικολογική αυτή καταστροφή ε, που είναι κυρίως πλωτά σκουπίδια από την Αλβανία και το Μαυροβούνιο τα οποία παρασύρονται προς τα κροατικά νησιά. Προσωπικά έχω απευθύνει έκκληση στην Κομισιόν για να προληφθεί αυτή η οικολογική καταστροφή παρά το ότι αυτές οι χώρες έχουν υπογράψει την ε, σύμβαση της Βαρκελόνης για την προστασία της, ε, του θαλασσίου περιβάλλοντος της Μεσογείου, ο αριθμός των ε, θαλασσίων αποβλήτων αυξάνεται. Αναμένω λοιπόν τη στρατηγική σας για τα πλαστικά την οποία ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, αλλά θεωρείται ότι μια πιο αποτελεσματική περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των γειτονικών χωρών που είναι και υποψήφιες πλέον είναι αναγκαία για να εφαρμοστούν καλύτερα οι περιβαλλοντικές πολιτικές. Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής αυστηρότερων κριτηρίων για το άνοιγμα και κλείσιμο κεφαλαίων ε, για το περιβάλλον. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σπανία. Κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, ήμουν εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την ιστορική συμφωνία στο Παρίσι το Δεκέμβριο για την COP21 το 2015 και μετά την COP23 όμως είδα προσωπικές σας δηλώσεις που δεν κινούνται προς την κατεύθυνση της δράσης μας, της κοινή μας δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Είπατε δημοσία ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι ένα μύ, ένας μύθος που προωθούν οι δυνάμεις της αριστεράς για να καταπολεμήσουν το κεφάλαιο της βιομηχανίας. Όχι κύριε Υπουργέ, ε, ο πλανήτης βρίσκεται σε κίνδυνο και εμείς θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που θα καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Ελπίζω λοιπόν αυτό το εξάμεινο να βάλετε κατά μέρος τις προσωπικές σας πεπιθήσεις και να προωθήσετε το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις κλιματικές αλλαγές. Η Βουλγαρική Προεδρία θα ε, προβάλλει μία υπουργική διάσκεψη για, την, ε, για τις κλιματικές αλλαγές σε συνέχεια της διάσκεψης που οργάνωσε πρόσφατα ο πρόεδρος Μακρόν, η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εδώ είμαι. Για αυτά τα οποία μας είπατε. Να αναφερθώ στρατηγική για τα πλαστικά. Πολύ σημαντική στρατηγική της Κομισιόν και είναι πολύ θετικό το ότι την καθορίζεται ως προτεραιότητα. Μπορώ να σας πω ότι προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με πολλούς βουλευτές να χαράξουμε μια τέτοια πολυετή στρατηγική. Αν πετύχει τον Απρίλιο, ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι ε, από κοινού. Μετά, συγκεκριμένα. Να αναφερθώ λίγο στις θάλασσες που με ενδιαφέρουν. Η Βουλγαρία βρέχεται από θάλασσα. Έχουμε την Διεθνή Διακυβέρνηση των Θαλασσών από την Κομισιόν και η υγεία των θαλασσών είναι ένα σημαντικό θέμα και για την κλιματική αλλαγή και για όλους μας. Το ερώτημα είναι, υπάρχει 1η Ιουνίου στο Μπουργκάς ε, οργανώνεται την Ευρωπαϊκή ημέρα των θαλασσών. Η ερώτησή μου λοιπόν, τι θα κάνετε ως Υπουργό Περιβάλλοντος. Έχετε κάποια πράγματα που θα θέσετε προστασία της βιοπικιλότητας ή ε, κλιματική αλλαγή ή κάτι άλλο. Ποιος είναι ο ρόλος σας. Αυτό θα με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι ως Υπουργός Περιβάλλοντος οπωσδήποτε και εσείς θα τοποθετηθείτε και θα είστε εκεί. Σας ευχαριστώ, κυρία Καμπεσού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ως προς τις ε, κλιματικές αλλαγές ε, ότι με σοκάρει κάπως η πρότασή σας ε, γιατί μιλάμε για κλικική οικονομία, για τα πλαστικά αλλά ως προς τις κλιματικές αλλαγές υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Είναι ένα μεγάλο λάθος και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης στην οποία αναφερθήκατε και εσείς. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο, μάλλον ποια είναι η θεώρησή μας ε, ως προς τις κλιματικές αλλαγές, γιατί ας πούμε όταν εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι ήταν διαφορετικές οι θεωρίες για την εξαφάνισή τους την κεντρική και ανατολική Ευρώπη υπάρχουν πολλές πυρκαγιές, το ίδιο και στη Νότιο Ευρώπη και χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό καταπολέμησης. Η Επιτροπή προέβαλε ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένας εύρωστος ε, μηχανισμός διότι όλα εξαρτώνται από τη γεωγραφική ζώνη. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι σε κάθε γεωγραφική ζώνη και για πρόληψη και για θεραπεία. Θα πρέπει λοιπόν μέσω και μακροπρόθεσμα να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπως τελευταίες πυρκαγιές που αντιμετωπίσαμε στην Πορτογαλία. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό το πλαίσιο διότι έχει μεγάλη σημασία να λάβουμε υπόψη το ΑΕΠ αυτής της γεωγραφικής ζώνης, μάλλον των γεωγραφικών ζωνών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμοφ, ευχαριστούμε που ήρθατε να μας αναπτύξετε σήμερα τους στόχους της Βουλγαρικής Προεδρίας στις ε, παρατηρήσεις σας τονίσατε ότι η Βουλγαρική Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στις προσπάθειες ε, για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Απέρα πέρα από τα προσωπικά σας προβλήματα με την κλιματική αλλαγή εκπροσωπείται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα με ενδιαφέρει λοιπόν ε, το εάν εργάζεστε προς την εξή κατεύθυνση να περιληφθούν στις σχετικές προσπάθειες της Ένωσης οι εκπομπές από την γεωργία. Γιατί είναι ένα ταμπού αυτή τη στιγμή. Οι εκπομπές ε, από την μαζική κτηνοτροφία είναι τόσο μεγάλες πια ώστε πρέπει να αντιδράσουμε και να μην κλείνουμε τα μάτια μόνο και μόνο επειδή είναι ένα ακαθόδες θέμα που αφορά την διατροφή μας. Τα παραγωγικά ζώα, ειδικά τα βοηδή, εκπέμπουν πολύ και χρειαζόμαστε μια προεδρία που θα τολμήσει να το κατονομάσει. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν έχετε το θάρρος ή όπως και οι προηγούμενοι συναδελφοί σας θα κάνετε την πάπια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Βόλκεν. Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ειλικρινά σοκάρομαι λίγο από την συζήτηση που ακούω. Δεν αρκεί να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει συνένεση για την κλιματική αλλαγή και να πούμε ότι αρκεί αυτό για Προεδρία του Συμβουλίου. Η πολιτική ατζέντα είναι ελάχιστη και θεωρώ ότι όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει επιστημονική συνένεση για την κλιματική αλλαγή και, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να επιτύχει κάτι ε, είναι νομίζω λανθασμένο να την αμφισβητούμε έτσι. Έχω μια ερώτηση για την οδηγία περί ποσίμων υδάτων ε, που αφορά και τους συναδέλφους. Ε, την αναμένουμε. Έχουμε ένα εκατομμύριο πολίτες ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν ε, καθαρό νερό, πόσιμο. Ξέρετε ότι η οδηγία αυτή βασίζεται στο δικαίωμα στο νερό, είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς και υπάρχουν δύο δυνατότητες που προτείνονται για το πώς ε, το ένα εκατομμύριο αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν πόσιμο νερό είτε μέσω μιας σύνδεσης ε, τρεχούμενου νερού είτε μέσω κάποιας άλλης δυνατότητας. Θα ήθελα να μάθω τι έχετε να μας πείτε. Η κυρία Κάδενμπαχ, τελευταία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Την επόμενη ερώτηση θα την περιμένετε μάλλον. Θα αναφερθώ οπωσδήποτε στο Πύρι. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή όπως μου λένε, δεν έχω πάει. Υπάρχει ανησυχία εκεί τον ΜΚΟ που φοβούνται ότι η ποιότητα αυτού του εθνικού δρυμού που είναι το οποίο παγκόσμιας κληρονομιάς ε, και έχει δύο περιοχές Natura 2000 ε, θα κινδυνεύσει από τα προγραμματιζόμενα έργα ανοικοδόμησης. Ε, τονίζεται συνεχώς ότι πρόκειται απλά για διόδους ε, και για τελεφερίκ. Αλλά βεβαίως ε, αυτό απαιτεί υποδομή και διάφορα άλλα πράγματα. Και μιλάμε για ένα 42% του πάρκου το οποίο θα είναι διαθέσιμο όπως μας λέτε για υδροδότηση στο μέλλον. Αυτό όμως σύμφωνα με την ε, βουλγαρική νομοθεσία επιτρέπεται μόνο για πόσιμο νερό. Ε, υπάρχει ένας φόβος λοιπόν εδώ. Εμείς θεωρούμε ότι ο τρόπος ε, που επιλέξατε στις 21 Δεκεμβρίου δεν συμφωνεί πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουμε και τη οδηγία αξιολόγησης του περιβάλλοντος. Θα ήθελα λοιπόν να μας απαντήσετε κάτι. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε εδώ ο κατάλογος, αλλά υπάρχει λίγος χρόνος. Αν λοιπόν θέλει κάποιος άλλος τον λόγο. Όχι. Το διάει μάλιστα, ωραία. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να απαντήσω πάλι με χρονολογική σειρά. Αλλά υπήρχαν και τέσσερις ερωτήσεις που ήταν παρόμοιες και θα τις απαντήσω μαζί. Κυρία Σουίτσα μίλησε για κυκλική οικονομία ως προτεραιότητα της Βουλγαρικής Προεδρίας. Στις 16 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το μίνι πακέτο, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, πριν από μια εβδομάδα. Οπότε το αναμέναμε. Η κυκλική οικονομία, μιλώντας ως πρόεδρος του Συμβουλίου, είναι ένας από τους κινητήρες, θα έλεγα, που ενθαρρύνει την οικοκαινοτομία. Θα δώσουμε προτεραιότητα στην στρατηγική για τα πλαστικά και θα ξεκινήσει και μια συζήτηση στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος τον Μάρτιο. Θα εστιαστεί η συζήτηση στο πώς θα αυξηθεί η ανακύκλωση ε, θα μειωθεί ο ενταφιασμός σε χωματερές και η απαντράκωση. Οπότε σκοπεύουμε να ευθύσουμε όπως είπα συμπεράσματα τον Ιούνιο και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στην Κομισιόν για το ποια μέτρα θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα ποια πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα και γρήγορα. Οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώ ε, πώς ε, επηρεάζονται αυτές οι νομοθεσίες περί χημικών και αποβλήτων τώρα. Κύριο Σπαρνιό. Ο κ. Καμποστρουής, ΕΚ και Βόλκεν μίλησαν για την κλιματική αλλαγή. θα τα συνοψίσω αυτά και μετά υπήρξε και μια ερώτηση για το νερό. Το θέμα της πολιτικής συνένεσης δεν πρέπει να το υποτιμάμε γιατί ε, δεν υπάρχει συνένεση στην επιστήμη αλλά υπάρχει στην πολιτική. Στην πολιτική η συνένεση είναι ένα βασικό μέσο για να επιτύχουμε τους ε, στόχους μας. Είναι πολύ σημαντικό όμως. Εάν δεν υπάρχει συνένεση οι στόχοι αυτοί θα έχουν αντιπάλους. Στην επιστήμη δεν μιλάμε για συνένεση γιατί όπως είπα η επιστήμη πάντα αναζητεί την αλήθεια. Υπάρχει αμφιβολία γιατί αν υπήρχε συνένεση δεν θα υπήρχε πρόοδος. Οπότε κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής ε, προεδρίας ε, θα, εργαζώ... θα εργαστούμε στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής συνένεσης των 28 και με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε θα διατηρηθεί αυτή η συνένεση. Δεν βλέπω λοιπόν λόγο ανησυχίας. Ο υπουργό ε, Περιβάλλοντος επίσης ε, προεδρεύω και του Συμβουλίου. Και στόχος μου είναι ακριβώς αυτή η συνένεση. Ο κ. Βέλκεν μίλησε για το πόσιμο νερό. Η απάντησή μου αυτή, ε, όπως είπα, αφορά και την ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συζήτησα λοιπόν αυτό το θέμα ε, και το ανέφερα και όταν μίλησα και για την ποιότητα του αέρα. Αλλά και το νερό είναι εξίσου σημαντικό. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πέντε προτεραιότητες ε, ταυτόχρονα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η υγεία και οτιδήποτε αφορά την υγεία. Οπότε θα υπάρχουν εξέλιξεις ε, όσον αφορά το νερό. Τώρα, υπήρχε ένα ερώτημα τη κυρία Καπεζών, Ρουίσα, για την πολιτική προστασία. Ως ε, πρόεδρος ε, θα φροντίσω να αναζητήσουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ε, προστασίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων και την δυνατότητα αντιμετώπισης θεομηνιών. Αντιλαμβανόμαστε την πολιτική σημασία τους, γι' αυτό θέλουμε να επιτύχουμε. Θεωρούμε ότι θα ανταποκριθούμε στις ε, προσδοκίες των πολιτών και θα υπάρχει γρηγορότερη αντίδραση ε, των μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Τώρα, η κυρία Μάισνερ. Α, όχι, όχι. Όχι απάντησα στην κυρία Μάισνερ ήδη. Λοιπόν, η κυρία Κάντενμπαχ. Ναι. Ζητώ συγγνώμη. Δεν απάντησα στην ερώτησή σας. Με ρωτήσετε για ένα ζήτημα εθνικό της ε, Βουλγαρίας, ε, το οποίο δεν αφορά βεβαίω ε, τον ρόλο μου εδώ πέρα σήμερα ως Προεδρεύον του Συμβουλίου. Αν θέλετε να σας απαντήσω μετά σε διμερές επίπεδο. Αλλά να σας πω για να μην πείτε ότι αποφεύγω την ερώτηση. Πρόκειται για μια προστατευμένη περιοχή υπό την προστασία της UNESCO. Είναι τουριστική ζώνη και ακριβώς μιλάμε μόνο για αυτήν την ε, ζώνη προστασίας. Το άλλο νούμερο, το 45% που αναφέρατε, χρησιμοποιείται για ε, πόσιμο νερό. Αυτό το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν είναι αντίθετο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μιλάμε για πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Ε, όλοι χρειάζονται καθαρό νερό. Δεν βλέπω λοιπόν εγώ κάποια αντίφαση εδώ πέρα. Ο Επιτροπός Βέλλα σε μία συνέντευξη είπε ότι δεν έχει παραβιαστεί ε, η βουλγαρική νομοθεσία ούτε και η ευρωπαϊκή βεβαίως και δεν νομίζω να παραβιάσουμε κάποιο νόμο βουλγαρικό ή ευρωπαϊκό. Μια στιγμή. Α, κυρία Μάισνερ, ζητώ συγγνώμη. Μιλήσατε ναι, για την ημέρα των θαλασσών, την εκδήλωση που θα γίνει στον Μπουργκάς 31 ε, Ιανουαρίου και το γεγονός ότι υπάρχουν σκουπίδια στη θάλασσα, υπάρχει ρήπανση. Ναι. Θα γίνει λοιπόν μια εκδήλωση Θέλουμε να είναι καθαρές οι θάλασσες. Έχουμε ένα έργο που γίνεται για τη χαρτογράφηση της Μαύρης Θάλασσας και πάλι υπό το Natura 2000. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά άμεσα την Βουλγαρία και θα ήθελα να απαντώ σε ερωτήσεις ως πρόεδρος του Συμβουλίου, εκπροσωπώντας και τις 28 για όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν, τα οποία βρέχονται από θάλασσες ή έχουν ε, σχέση με την κατάσταση των ε, θαλασσών. Αυτό βέβαια είναι και θέμα οικονομίας. Μόνο η ισορροπία μεταξύ οικονομίας και περιβάλλοντος θα μας οδηγήσει σε ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Με χαρά μου λοιπόν ε, να σας προσκαλέσω, αν μπορείτε να έρθετε, στις 31 ε, του μηνός, στο Μπουργκάς, όλοι σας, όσοι θέλετε. Πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε με τους ευρωβουλευτές θα είναι χαρά μας λοιπόν να σας φιλοξενήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για τις πληροφορίες, τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις μας. Ε, χαιρόμαστε και εκτιμούμε για το γεγονός ότι παρευρεθήκατε εδώ μεταξύ μας. Σας ευχαριστούμε και για την πρόσκληση και πολλοί από εμάς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τιμήσουμε την Βουλγαρική Προεδρία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κλιματικές αλλαγές. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία για το επόμενο εξάμεινο.